φυλακή και παραβιάζοντας την νομοθεσία της χώρας δεν τους επιτρέπουν να επισκεφθούν την κυρία Τιμοσέγκο, η κόρη της και ο δικηγόρος. Ευχαριστώ ε, για την ανακοίνωση αυτή που είναι πολύ λυπηρή και δείχνει πόσο έχει κλιμακωθεί η κατάσταση στην Ουκρανία και πόσο σημαντική θα είναι η επόμενη διαδικασία και από πλευράς Κοινοβουλίου με την έγκριση του ψηφίσματός μας. Ερχόμαστε λοιπόν στις ψηφοφορίες σύμφωνα με την ημέρα διάταξη. Έκθεση Τάιν. Μία είναι η ψηφοφορία και μάλιστα ονομαστική αρχίζει τώρα. Εγκρίνεται. Η κυρία Συγήτρια ζητεί το λόγο, παρακαλώ. Η κυρία Τέν. Αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σε συμφωνία με όλες τις πολιτικές ομάδες ζητώ αναβολή της τελικής ψηφοφορίας για το νομοθετικό ψήφισμα. Η ερχόμενη ελληνική προεδρία ε, θέλει την πρόταση του Κοινοβουλίου να τη συζητήσει. Με εξέπληξε αυτό ε, για τον αριθμό των δικαστών ε,